Το επόμενο είναι επεξηγήσει ψήφου. Να σα πληροφορήσω ότι έχουμε λάβει πολλές, ε, πολλά αιτήματα για επεξηγήσει ε, ψήφου. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίαση το αργότερο στις 3 ε, παρατέταρτο ούτω ώστε να ετοιμάσουν οι υπηρεσίε το επόμενο τμήμα συνεδριάσεις. Οι επεξηγήσεις ψήφου λοιπόν που δεν θα γίνουν τώρα θα έχουν κάποιο χρονικό περιθώριο, θα δοθεί αύριο.